Ανατολή, εγγυόμενη τα ανθρώπινα δικαιώματα, χωρί όμω να λυγίζει μπροστά στην υπεροψία, μπροστά στους εκβιασμούς και μπροστά στι ρητέ απειλέ του Ερντογάν ότι θα μας κατακλείσει με 3,6 εκατομμύρια μετανάστες. Όταν όμως αρχίζουμε και μιλάμε μόνο για κυρώσεις, όταν ε, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ουσιαστικά ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που χρηματοδότησε την Άγκυρα μέσω διαφόρων μέσων, όπως για παράδειγμα η προταξιακή βοήθεια, οι χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η, η όλη υποστήριξη που δόθηκε για τους πρόσφυγες στην Τουρκία. Τώρα λοιπόν, περισσότερο από ποτέ, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι θα πρέπει να σταματήσει η διαδικασία προσχώρησης Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια ενδεχόμενη προσχώρησή της θα οδηγούσε στην Ισλαμοποίηση της Υπήρου μας και ουσιαστικά οι χριστιανοί θα γινόταν μια πολύ μικρή εκδιωκόμενη μειονότητα όπως ακριβώς γίνεται τώρα στη Συρία. Ευχαριστώ. Έληξε ο χρόνος σας κυρία μου. Έχω κλείσει το μικρόφωνο σας, άρα κανείς δεν σας ακούει. Και τώρα ο επόμενος ομιλητής για ένα λεπτό, ο κύριος Χριστοφόρου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η εισβολή τη Τουρκία στη Συρία αποτελεί έναν ιδεχθέ έγκλημα, έγκλημα κατά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τη Ευρώπη και κατά τη ανθρωπότητα. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή είναι η ώρα να τελειώσουν τα λόγια στην ευρωπαϊκή ένωση και να αναλάβουμε δράση. μηδενική ανοχή στην τουρκία η οποία αυτή τη στιγμή δεν επιτίθεται απλά και μόνο στους Κούρδους. Επιτίθεται ενάντια στην ανθρωπότητα γιατί οι Κούρδοι ήταν αυτοί που αποτέλεσαν την ασπίδα για τη διάλυση του ISIS για να κοιμάται η Ευρώπη ήσυχη και η Ευρώπη αυτή τη στιγμή ουσιαστικά με την ανοχή τη κατατάσσεται σε αυτούς που θα θεωρηθούν συνένοχους για αυτόν το ιστορικό εγκληματικό λάθος ενάντια στην ανθρωπότητα. Η Τουρκία επαναλαμβάνει αυτό το 1915 ήταν η εξόντωση των Αρμενίων, το 1918 των Ελλήνων του Πόντου, το 1922 των Ελλήνων της Μύρνης, το 1955 της Κωνσταντινούπολης, το 1974 της πατρίδας μου της Κύπρου. Πέρσι ήταν το Ανφρίβ, φέτος είναι η γενοκτονία των Κούρδων. Δεν πρέπει να περιμένουμε άλλο. Θεωρώ τον εαυτό μου ότι είμαι περήφανο Ευρωπαίος, όμω νιώθω ντροπή όταν με ευρωπαϊκά όπλα οι Τούρκοι επιτίθενται στου Κούρδους και όταν ακόμα δεν λάβαμε αποφασιστικά μέτρα για να σταματήσουμε αυτή την εισβολή τη Τουρκία. Η κυρία Φαγιόν, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Στη Βόρεια Συρία υπάρχει μια πολύ αδύναμη κατάπαυση του πυρός, την οποία μπορεί να διακόψει όποτε θέλει ο Ερντογάν. Η έλλειψη ενότητας στην Ευρώπη του επιτρέπει να κάνει ό,τι θέλει. Είναι μια παραβίαση του διεθνούς δικαίου και οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να καταλήξουν σε κοινή θέση. Πρέπει να σταματήσουν οι πωλήσει όπλων προς την Τουρκία και να επιβληθούν οικονομικές κυρώσεις. Έτσι θα μπορέσουμε να πιέσουμε την Άγκυρα. Μόνο έτσι. Το θέμα της Τουρκίας δεν θα επιληθεί ακόμη και αν ε, αποσύρουν τα στρατεύματά τους από τη Βόρεια Συρία. Το κουρδικό θα συνεχιστεί να είναι θέμα. Να μην ξεχνάμε λοιπόν τις σχέσεις των Κούρδων με τον Ασάντ. Ακόμη και αν σταματήσουν οι επιθέσεις της Τουρκίας θα είναι πάντα πυρτιδαποθήκη αυτή η περιοχή όπου θα υπάρχουν δεινά για τους λαούς και ροές προσφύγων. Είναι ντροπή η πορεία της ανθρωπότητας αυτή τη στιγμή. Η κυρία Παγαθορτουντούα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Με πολύ προσοχή άκουσα αυτή την ε, μακρά συζήτηση. Είμαστε απογοητευμένοι. Αλλά ε, δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε και τόσο φοβισμένοι. Φοβισμένοι είναι αυτοί οι οποίοι βλέπουν τις βόμβες να πέφτουν επάνω τους. Να μην ε, υποκρινόμεθα ότι δεν ξέραμε ότι θα καταλήψουν την περιοχή οι ΗΠΑ. Ξέραμε ότι θα επιτεθεί η Τουρκία. Το ξέραμε. Ότι θα δραπέτευαν επικίνδυνοι μαχητές ότι θα δημιουργηθεί μια κλιμάκωση αναβίωσης του Ισλαμικού κράτους της τρομοκρατίας. Τα ξέραμε, μας είχαν προειδοποιήσει όλοι. Χάσαμε μια ευκαιρία νωρίτερα πριν από την απόσυρση των ΗΠΑ. Έπρεπε να έχουμε δράσει με ένα διεθνές ποινικό δικαστήριο για να αποφύγουμε την ασυδοσία όλων αυτών, για να ε, κάνουμε κάτι για τους ανήλικους ε, που ζουν σε αυτή την περιοχή και που είναι πολίτες μας. Εμπορικά παίζουμε ένα ρόλο, πολιτικά όχι. Κοιτάξτε, σε έναν ε, παγκοσμιμένο κόσμο τέτοιε σειράξει μα επηρεάζουν πάντα. Σίγουρα θα μα επηρεάσουν. Εμεί προσπαθούμε ακόμη να αντιμετωπίσουμε μια μεταναστευτική κρίση που είναι επίπτωση αυτών των συγκρούσεων. Λοιπόν, εάν δεν σταματήσουν αυτέ οι αντιθέσει τη πολιτική μα, αν δεν έχουμε μια πολιτική ασφάλεια και άμυνα, δεν θα επιτύχουμε τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Ένα λεπτό. Ο κύριος Αλεξάνδρου Φεγιορτάνου. Ευχαριστώ. Η κατάσταση άλλαξε χθες. Ο Πούτιν και ο Ερντογάν πήραν αυτό που ήθελαν. Ο Πασάρα Λασάντ συμφωνεί παρόλο που είναι ένας από τους βασικούς ε, ενόχους για αυτή την κατάσταση. Η πολιτική της Τουρκίας δεν είναι απλώς κατά των Τούρκων αντικουρδική, είναι αντιευρωπαϊκή. Αντίκειται στις θέσεις μας. Πραγματικά θα πρέπει να έχουμε σοβαρές ανησυχίες για την διαδικασία αυτή που έχει προκύψει μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας. Δεν είναι μία, ένα απλό διπλωματικό φλερτ. Είναι μια πιο επικίνδυνη διαδικασία. Μπορούμε να προσφέρουμε λύσεις αυτό. Μπορούμε να δώσουμε ένα όραμα σχετικά με το πώς θα επιληθεί το πρόβλημα συμπεριλαμβανομένου και του κουρδικού ζητήματος. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα υποστηρίζουμε τους αριστεριστές, ε, τους ε, εθνικιστές ε, και όλους αυτούς που λειτουργούν μέσα στο, στην επικράτεια αυτή. Για ένα λεπτό, ο κύριος Χαϊναλούμα. Ε, κυρία Πρόεδρε, επιδρομή των Τούρκων είναι κατά του διεθνούς δικαίου. Δεν μπορούμε να την αποδεχτούμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς έχει παραμείνει ε, στο παρασκήνιο, απλώς να παρακολουθεί, ενώ η Τουρκία, οι Ηνωμένες η Ρωσία, ακόμα και η Ιράν οργανώνουν τα πράγματα στην περιοχή. Τα συριακά πετρέλαια έχουν περισσότερους, ε, έχουν περισσότερους να τους προστατεύουν και περισσότερα δικαιώματα από ότι οι Κούρδοι. Οι Κούρδοι στους οποίους χρωστάμε τόσα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν πρέπει να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα. Περιμένουμε από το Συμβούλιο την είπατε εκπρόσωπο για την Κομισιόν πιο αποφασιστικές δράσεις ώστε να δοθεί ένα τέρμα σε αυτή την τραγωδία και η Τουρκία να κατανοήσει τα όρια των επιχειρήσεών της. Αυτό σημαίνει αποφασιστική δράση ε, και μια ευρωπαϊκή ε, πολιτική ακόμα και με ένα εμπάργκο όπλων. Ευχαριστούμε για ένα λεπτό κύριος ε, Γκρούντλερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αυτός ο νέος πόλεμος στα βόρεια της Συρίας με πρωτοβουλία της Τουρκίας είναι παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Είναι απόφαση ε, η οποία δυστυχώς εκτοπίζει 200.000 ανθρώπου, 70.000 παιδιά και έχουμε και ε, τόσους ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους. Δεν είναι ένας πόλεμος κατά των τρομοκρατών, αλλά κατά του λαού, του λαού της, των Κούρδων, ε, που οι περισσότεροι από αυτούς ζουν σε ειρήνη και ελεύθερη. Είμαστε πολύ πιο δυνατοί ε, όταν είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον και όχι όταν είμαστε ο ένας κατά τον άλλον. Αυτό το είπε ο κύριος Ερδογάν. Ε, τα 30 χιλιόμετρα ζώνης ασφαλείας ε, που αυτός ε, με στρατιωτική πυγμή επιβάλλει είναι ακριβώς για αυτόν ένα εργαλείο ώστε να βάλει εκεί τους πρόσφυγες που λέει ότι θα πάνε εθελοντικά. Όμως θέλει να δεν λαμβάνει υπόψη το συμφέρον των ανθρώπων αυτών. Ο γολγοθάς αυτών των ανθρώπων δυστυχώς δεν έχει ακόμα τελειώσει. Ευχαριστούμε ο κύριος Λέγκα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι πλέον πέραν πάσης αμφιβολίας για όλους μας ότι ο Ερντογάν δεν ανήκει σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση και επεμβαίνοντας στη Συρία και χρησιμοποιώντας την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ως πρόσχημα, ουσιαστικά κατέστησε απολύτως σαφές ότι δεν ακολουθεί τους κανόνες της διεθνούς κοινότητος, όπως ακριβώς γίνεται και με την κατοχή της Κύπρου, όπως γίνεται και με την παραβίαση του ελληνικού φύρ, όπως γίνεται με τις γεωτρήσεις στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να καταφέρουμε να προστατεύσουμε και τους Κούρδους και τους Χριστιανούς, γιατί και αυτοί απειλούνται. Ο Ερντογάν έχει καταδείξει πλέον ξεκάθαρα ότι μισεί όλες τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ερντογάν μισεί τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωή, μισεί τη δημοκρατία, τις θεμελιώδει ελευθερίε, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τι ελευθερίε μα και το κράτο δικαίου. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η Τουρκία του Ερντογάν να νίκει ποτέ στο μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα πρέπει αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση να τερματίσει επιτέλου τι ενταξιακέ διαπραγματεύσει με την Τουρκία. Σα ευχαριστώ. Κύριο Σάρακοβα, έχει τώρα το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι περισσότεροι εξ ημών ενδεχομένω να έχουμε διαβάσει το βιβλίο το οποίο ονομάζεται οι 40 μέρε του Μουζαντάχ, το οποίο γράφτηκε τον προηγούμενο αιώνα. Έχουμε την περιγραφή μιας απέσια γενοκτονία, η οποία φαίνεται να επαναλαμβάνεται εκείνη τη στιγμή και εμεί δεν μπορούμε να σιωπούμε. Είναι απαράδεκτο μια κυβέρνηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, και αναφέρομαι στην Ουγγρική κυβέρνηση να έρχεται και να υποστηρίζει ένα αυταρχικό ολοκληρωτικό καθεστώ το οποίο έχει κηρύξει πόλεμο κατά των Κούρδων τη Συρίας και το οποίο τελικά αποστεθεροποιεί όλη την περιοχή και δημιουργεί μια ανθρωπιστική κρίση. Α πούμε τα πράγματα ξεκάθαρα. Ο Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίο θεωρεί ότι οι πρόσφυγε είναι εχθροί και που μα απειλεί με αυτού έχει αρχίσει αρχίσει τώρα να υποστηρίζει μία επέμβαση η οποία έχει εκτοπίσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Από την άλλη, ο τρόπος με τον οποίο εκτιλήσεται η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαράδεκτη. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να επιτρέψουμε σε πολιτικούς που δεν έχουν κανένα ηθικό έρισμα να εκπροσωπούν από κοινού την εξωτερική και διπλωματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώ καλό το Συμβούλιο να λάβει επιτέλους συγκεκριμένε αποφάσεις με ειδική πλειοψηφία και όχι μαμοφωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκρόισε, ένα λεπτό. Η επέμβαση στη Συρία είναι μία από τις χειρότερες ε, παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων αυτού του αιώνα αλλά αυτές πρέπει να είναι η βάση του σημερινού κόσμου. Και αυτή η επίθεση γίνεται από ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Και οι διάφορες πολιτοφυλακέ οι οποίες ε, συμμετέχουν διαπράττουν τι χειρότερες ε, θηριωδίε. Ο Ερντοάν λέει ότι θέλει να αποκαταστήσει την ειρήνη στην περιοχή, αλλά να μην είμαστε αφελεί. Η συνάντηση στο Σότσι αποδεικνύει τι θέλουν. Είναι σίγουρα η επιβολή των γεωστρατηγικών συμφερόντων ε, της Τουρκίας χωρίς κανένα όριο. Δεν είναι καταπολέμηση της ε, τρομοκρατίας, γιατί αλλιώ η Τουρκία δεν θα επιτίθεται στους Κούρδους που είναι οι μόνοι που πολέμησαν με τα όπλα στο χέρι το Ισλαμικό κράτος. Οι απειλές του Ερντοάν και οι εκβιασμοί προς την Ευρώπη με περισσότερους πρόσφυγες είναι σαφής ενδείξει ότι θέλει να χρησιμοποιήσει τα δεινά που υφίστανται εκατοντάδε χιλιάδε άτομα για να εξυπηρετήσει του σκοπού του. Πρέπει να είμαστε στο ύψο αυτή τη πρόκληση. Η Ένωση πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει τι εξελίξει, να πιέζει την Τουρκία. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε. Δεν το ξέρω. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Μάντλ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μία παροιμία λέει ότι το πρώτο θύμα σε κάθε πόλεμο είναι η αλήθεια και ο τίτλος αυτής της, ε, το, αυτής της ε, ε, επίθεσης των Τούρκων «Πηγή ειρήνης» είναι πραγματικά τεράστιο ψέμα. Είναι πηγή θηριωδιών, βίας και εκτοπισμού. Η Τουρκία δεν έχει καμία εκτίμηση για τις ευρωπαϊκές αξίες. Άρα δεν πρέπει να έχει καθεστώς υποψήφιας χώρας. Πρέπει να τις αφαιρεθεί. Είναι, μα είναι παράλογο, συνάδελφοι μια πολύ μικρή και άθλια μειοψηφία της, ε, στο Συμβούλιο παρεμποδίζει τη χορήγηση καθεστώτος ε, υποψηφίου μέλους στην ε, Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία που έχουν κάνει τόσο πολλά, ενώ η Τουρκία εξακολουθεί να το έχει. Θα πρέπει οπωσδήποτε να πιέσουμε την ίδια δύναμη ευρωπαϊκή οικονομία μέσω αναστολής της Τελειωνιακής Ένωσης. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο μισός ε, τουρκικός πληθυσμός δεν στηρίζει το καθεστώς, αλλά το καθεστώς θα πρέπει να δράσει ψύχρεμα και αν πιέσουμε την οικονομία θα το κάνει. Εμείς πρέπει να εκφράσουμε τη φωνή των Ευρωπαίων όλων να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κ. Ανδρουλάκης. Ένα λεπτό. Ενάμιση περίπου χρόνο σε αυτή την αίθουσα συζητούσαμε πάλι για την τουρκική εισβολή στο Αφρίν από τη συγκεκριμένη επιχείρηση το μόνο που άλλαξε είναι το όνομα. Από τον κλάδο ελέας περάσαμε στην πηγή ειρήνης. Ας μιλήσουμε όμως καθαρά. Ο Ερντογάν από πρωταγωνιστή στο παρασκήνιο σταθεροποίηση της Συρίας πλέον και με την ανοχή της διεθνούς κοινότητας και των μεγάλων γεωπολιτικών παιχτών της περιοχής χτυπάει τους Κούρδους. Αυτούς που αντιστάθηκαν στο Ισλαμικό κράτο και τα εγκλήματα κατά τη ανθρωπότητα που προκάλεσε. Μετά από 8 χρόνια ματηρού εμφυλίου, η τουρκική εισβολή αποτελεί πηγή αίματος και ανθρώπινης κρίσης και όχι πηγή ειρήνης όπως ηρωνικά τη βάφησε ο κύριο ερντογάν ο οποίος δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο όσο και αν εμείς φωνάζουμε. γι' αυτό τώρα χρειάζονται πραγματικές κυρώσεις. ένα άμεσο πανευρωπαϊκό εμπάργκο όπλων που δεν θα περιορίζεται σε νέες παραγγελίες αλλά θα τερματίζει την παράδοση όπλων από όλα τα κράτη μέλη άμεσα με στοχευμένες κυρώσεις σε όσους έχουν την ευθύνη για την εισβολή και βέβαια και σε εμπορικές κυρώσεις που θα αποδεικνύουν ότι η ευρώπη εννοεί αυτά που λέει. Ο για ένα λεπτό το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, η απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από την βορειοανατολική Συρία ήταν ένα γεγονός που ουσιαστικά εξέθεσε σε πολύ μεγάλο κίνδυνο τους Κούρδους και τους Χριστιανούς της Συρίας. Και είπε μάλιστα ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι στα πλαίσια της υπέρτατης σύνεσης και σοφίας του πήρε την κατάλληλη απόφαση, η οποία προφανώς δεν λειτουργεί στην πράξη. Δυστυχώς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και κυρίως το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων έλαβε μια απόφαση η οποία υπολείπεται πάρα πολύ του επίπεδου αντίδραση που θα πρέπει να έχουμε εδώ πέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε περισσότερε εξηγήσει. Νομίζω ότι οι αποφάσει που έλαβε το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων δεν βοηθάνε καθόλου του Κούρδου. Έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου να καταφέρουμε να λάβουμε συγκεκριμένε στοχευμένε οικονομικέ εμπορικέ κυρώσει. Θα πρέπει να σταματήσουμε τι εμπορικέ συναλλαγέ με τη χώρα αυτή. Οι Κούρδοι και οι Χριστιανοί εμπράκτο θα πρέπει να υποστηριχθούν οπουδήποτε και αν βρίσκονται. Σας ευχαριστούμε κυρία Μπάρντι για ένα λεπτό. Νομίζω ότι ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση για αυτή την ε, περιοχή. Πρέπει να είναι πολιτική η λύση μέσα από τα Ηνωμένα Έθνη που δεν έχουν καν αναφερθεί σε αυτή τη συζήτηση σήμερα. Σήμερα βιώνουμε μια ε, τουρκική εισβολή με την άδεια της ε, Ρωσίας. Οι δημοκρατικές δυνάμεις των Κούρδων που είναι οι καλύτεροι σύμμαχοι της διεθνούς κοινότητας έχουν μείνει ξεκρασμένοι δεν ε, De facto, λοιπόν, όλα αυτά γίνονται στη Σύρια, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μεγάλος παίχτης σε αυτή την περιφέρεια. Πέρασε ο χρόνος ε, και δεν έχουμε και τις ικανότητες ε, και βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δράσει, αλλά δεν έχει τις ικανότητες. Υπάρχουν οικονομικές κυρώσεις, το σταμάτημα των παραδόσεων όπλων. Αυτά θα πρέπει να συνεχίσουν και να μην εκβιαζόμαστε με, με ζητήματα που αφορούν σε πρόσφυγες. Thank you. Ευχαριστώ κύριο Ζόιντο Αλβάρης για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Στη σημερινή συζήτηση κατέστη σαφές ότι η στρατιωτική επέμβαση της Τουρκίας έχει δραματικές επιπτώσεις στο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό τομέα. Εγώ θέλω να τονίσω το θέμα της απελευθέρωσης χιλιάδων μαχητών του Άισις με ευρωπαϊκά διαβατήρια. Μπορούν να επανέλθουν στην Ευρώπη. Άρα θα έχουμε προβλήματα ασφάλειας παντού στην Ένωση. Θα είναι ανεξέλεγκτοι. Θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Στην Ισπανία έχουμε υποστεί την τρομοκρατία της ΕΤΑ για δεκαετίες με χιλιάδες θύματα. Αλλά χάρη στην εργασία των δυνάμεων ασφαλείας εκριζώθηκαν. Χάρη στη στήριξη και της ισπανικής κοινωνίας και την λειτουργία του κράτους δικαίου. Γι' αυτό θεωρούμε ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας μπορεί να γίνει μόνο με μια πολιτική εξωτερικών και άμυνας από πλευράς της Ένωσης πιο φιλόδοξη, πιο πλήρη. Μόνο έτσι θα αποφύγουμε την ανεξέλεγκτη δράση των μαχητών του Ισλαμικού κράτους. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λόπεθ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα πρέπει να στείλουμε ένα κατηγορηματικό μήνυμα ότι απορρίπτουμε και καταδικάζουμε την τουρκική επέμβαση που παραβιάζει το διεθνέ δίκαιο, τους ε, διεθνεί θεσμού, τα Ηνωμένα Έθνη, το ΝΑΤΟ, έχει πολύ σοβαρές ανθρωπιστικές ε, συνέπειες, αποσταθεροποιεί μια περιοχή, επαναφέρει τον πόλεμο σε μια περιοχή που έχει ήδη θυγεί και μετατοπίζει πληθυσμούς. Όλα αυτά γίνονται με την συνενοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Και τα θύματα είναι οι Κούρδοι, οι σύμμαχοί μα μέχρι τώρα στην καταπολέμηση και την εκρίζωση του Ισλαμικού κράτους και σαφή κέρδη και για τον Άσαντ και τον Πούτιν στην περιοχή. Άρα πρέπει να καταδικάσουμε την επέμβαση και να είμαστε κατηγορηματικοί να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουν διάθεσή μας. Απαγόρευση πώληση όπλων. Να χρησιμοποιήσουμε και την αγορά μας από την οποία να ωφελείται η Τουρκία και να πάρουμε αποφάσεις για την διαδικασία ένταξης. Δεν έχει έννοια η διαδικασία αυτή για την Τουρκία πλέον. Ο κύριος Μπίλτσικ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπόθηκε πολλές φορές, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το επαναλάβουμε. Η τουρκική επέμβαση στη βροντολική Συρία απειλεί τη σταθερότητα όλης της περιφέρειας. Ενισχύει ουσιαστικά όσους θέλουν να δημιουργήσουν μια νέα διένεξη στη Μέση Ανατολή. Είναι προς το δικό μας ζωτικό συμφέρον τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των κρατών μελών να πολεμήσουμε για την εδαφική ακαιρεότητα τη Συρία. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε η, να ξανασχεδιαστούν με τη στρατιωτική πυγμή τα σύνορα. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε αυτούς που είναι υπεύθυνοι για την προσάρτηση, την παράνομη της Κρυμαίας να κάνουν κάτι αντίστοιχο αυτή τη στιγμή στη Συρία. Επομένως χρειαζόμαστε μπάρκο όπλων, χρειαζόμαστε οικονομικές κυρώσεις, χρειαζόμαστε αναστολή των να διαπραγματεύσεων με την Τουρκία. Αυτά είναι τα, μέτρα τα οποία μπορούμε να αναλάβουμε άμεσα, εδώ και τώρα. Εν γέννη όμως θα πρέπει να δίνουμε μάχη και για τις ευρωπαϊκές αξίες στην άμεση γειτονία μας. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να επηρεάζουν τα πράγματα οι Ρώσοι και οι Τούρκοι που έχουν φτάσει πλέον στην άμεση γειτονία μας. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μαγιορίνο έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ο Έρντογαν προχώρησε στρατική επέμβαση σε πραγματική πράξη πολέμου. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και γι' αυτό το λόγο δική μα ανταπόκριση θα πρέπει να είναι πάρα πολύ σκληρή. Μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση δυσκολευόταν πάρα πολύ να μιλήσει με μια ξεκάθαρη και νέα φωνή. Νομίζω ότι δεν χρειαζόμαστε πλέον γενικέ αποδοκιμασίε. Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένε πράξει. Η στρατιωτική επέμβαση τη Τουρκία είναι μια πράξη ε, που θα πρέπει να τιμωρηθεί με συγκεκριμένες οικονομικές κυρώσεις με το εμπάρκο των όπλων. Θα πρέπει να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να καταφέρουμε να προστατεύσουμε τους άνδρες και τις γυναίκες του κουρδικού πληθυσμού. Να καταφέρουμε επιτόπου να συνδράμουμε τον πληθυσμό αυτό τον κουρδικό προς τον οποίο πρέπει να δείξουμε μια τεράστια αλληλεγγύη. Ένας πληθυσμός που χρησιμοποιήθηκε αρχικά για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και έπειτα εντελώς επονίδης εγκαταλείψαμε τους ανθρώπους αυτούς, τους γυρίσαμε την πλάτη. Α μην λυγίσουμε επίση απέναντι στην απειλή του Ερντογάν για του πρόσφυγε. Και για του πρόσφυγε όμω αυτού θα πρέπει να σταματήσει ο πόλεμο αυτό και θα πρέπει να αποσυρθούν από τη Συρία άμεσα τα τουρκικά στρατεύματα. Ο κύριο Κεφαλογιάννη έχει το λόγο για ένα λεπτό. Η Τουρκία με το πρόσχημα ότι οι Κούρδοι που κατοικούν στη Συρία είναι συλλήβδιν τρομοκράτες εισέβαλε στη χώρα αυτή και προχωρά σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στο συριακό έδαφος με θύματα αμάχους και αθώα παιδιά. Είναι η ίδια χώρα που το 1974 με ένα παρόμοιο πρόσχημα εισέβαλε στην Κυπριακή Δημοκρατία και από τότε έχει υπό την κατοχή της το 40% του νησιού. Προσυπογράφουμε όλοι μας την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που καταδικάζει απερίφραστα τη στρατιωτική επέμβαση που προκαλεί εκατοντάδες ανθρώπινα θύματα, θέτει σε κίνδυνο τον αγώνα εναντίον του ISIS και γύρει σοβαρή απειλή στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Καταδικάζομαι την επίθεση στη Συρία της Τουρκίας, χωρίς αστερίσκους και χωρίς υποσημειώσεις σας ευχαριστώ κυρία πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Μάρκες. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το 2017 η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε έναν μηχανισμό, μια διευκόλυνση. Στόχος ήταν να βοηθήσουμε τα 3,6 εκατομμύρια σύρων προσφύγων που είναι 0,7 του πληθυσμού της Ένωσης των 28 και είναι κατεστημένη στην Τουρκία. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το κλείσμα των συνόρων μας, η περιοριστική ερμηνεία της συμφωνίας του Δουβλίνου προκάλεσε ορισμένα κράτη-μέλη να συνεχίσουν να μπλοκάρουν την αλλαγή. Η έλλειψη αλληλεγγύης από πλευράς κάποιων κρατών μελών της Ένωσης έναντι των υπολείπων που υποδέχτηκαν το μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων. Όλα αυτά κατέστησαν αναγκαίο αυτό το μηχανισμό Ένωση Τουρκία. Και έκτοτε μα εκβιάζει συστηματικά η Τουρκία. Μα απειλεί πάντα ότι θα ανοίξει τη στρόφιγγα. Και βλέπουμε ότι και τώρα το κάνει. Εάν η Τουρκία για ε, κατανοητούς λόγους ασφαλείας ξεκινάει τέτοιες απαράδεκτες υποθέσεις δεν είναι δυνατόν να θεωρήσουμε ότι το ένα προκύπτει εκ του άλλου. Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση. Πρέπει να μιλήσουμε με μία φωνή, να κινητοποιήσουμε όλε τι δυνατότητε επιρροή, να συνεργαστούμε με τα Ηνωμένα Έθνη, ούτω ώστε να υπάρξει η ειρήνη σε αυτή την περιοχή που είναι θύμα τόσων ε, θηριωδίων. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Σον Κέλλη, ένα λεπτό. Κοιτάξτε, πολύ συχνά, όχι δεν είναι συχνά, που όλες οι πλευρές του Κοινοβουλίου συμφωνούν. Σήμερα συμφωνούμε όλοι καταδικάζοντας ε, αυτά που κάνει η Τουρκία στη Βόρεια Συρία. Είναι σαφές ότι όλοι συμφωνούμε και για τα αίτια της. Είναι η απόσυρση από τον Τραμπ των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων. Ε, και αυτό είναι συνεπές με την όλη του εικόνα. Και ποιες είναι οι επιπτώσεις όλα αυτά τα δεινά. Αυτά τα πράγματα τα εφίστανται οι Κούρδοι εδώ και γενναίες. Ούτως ή άλλως τώρα έχουμε το νέο κύμα προσφύγων, 230.000 ε, άτομα έχουν ε, μετατοπιστεί και το Ισλαμικό κράτο ε, ανακτά τις δυνάμεις του. Πρέπει λοιπόν να απαγορευτούν οι εξαγωγές όπλων προς την Τουρκία. Πρέπει να επανεξετάσουμε την οικονομική βοήθεια που δίναμε στην Τουρκία. Πρέπει να υπάρξει πολιτική λύση υπό την αιγίδα των ΗΠΑ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, είναι καλό που μπορούμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σχέδιο ψηφίσματος ε, το καθιστά ξεκάθαρο. Η Τουρκία ε, πρέπει να γνωρίζει ότι η υποστήριξή μας δεν είναι χωρίς όρους. Η Τουρκία υποτίθεται ότι θα ε, συνεχίσει να εργάζεται ως προς την ε, τήρηση των ευρωπαϊκών ε, στάνταρ. Αυτό όμως είναι ένα ξυπνητήρι για μας. Είναι μία αφύπνιση ότι η στρατηγική μας, η σωστή μεταναστευτική πολιτική είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει μια καλή λύση ειρήνης στην περιοχή και να μην μπαίνουν ε, οι στρατοί των άλλων χωρών ε, να αποσταθεροποιούν τις χώρες ε, και να μην σκοτώνονται άνθρωποι. Ευχαριστούμε κύριε Σπούρλας για ένα λεπτό. Ευχαριστούμε κύριο Σπούρλας ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κλείσαμε τα μάτια μπροστά σε ένα έγκλημα. Αφήσαμε τους ανθρώπους που πολέμησαν τον Άισις έρμεως στα χέρια της Τουρκίας. Και συζητάμε εδώ σήμερα στην Ευρώπη αν θα πρέπει να πάρουμε και πότε μέτρα να σας θυμίσω ότι πριν από 45 χρόνια η τουρκία ονόμασε ειρηνευτική επιχείρηση την εισβολή στην πατρίδα μου. 45 χρόνια μετά έχουμε ακόμα 200.000 χιλιάδες πρόσφυγες ξεσπιτωμένους και αγνοωμένους. και όπως τότε πριν από 45 χρόνια σιωπήσαμε η διεθνής κοινότητα σιώπησε και άφησε την τουρκία να ολοκληρώσει το έγκλημά της στην κύπρο. έτσι και σήμερα σιωπά και πάλι. συρία 2019 κύπρος 1974. Ο θήτης παραμένει ο ίδιος, παραμένει ατιμόρυτος. Και οι δικές μας ευθύνες τεράστιες και η Ευρώπη απούσα. Θα μας κρίνει η ιστορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βέντλα, ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, μιλάμε σήμερα για την παράνομη επιχείρηση της Τουρκίας στη Βόρεια Συρία και τις συνέπειες. Η κατάσταση εδώ και χρόνια είναι, είναι ε, δυσάρεστη ε, μετά από την, ε, τις πρόσφατες εξελίξεις με τον προφανή ρόλο Ρωσίας αλλά και του Άσαντ. Θα ήθελα να παρουσιάσω τα αιτήματα του ΕΛΚ στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δημιουργήσουμε ε, Συμβούλιο Άμυνας και να μπορούμε πρωτοβουλίες όπως της Γερμανίας για παράδειγμα να τις αντιμετωπίζουμε άμεσα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να μπορούμε να δρούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η απαράδεκτη ε, ενέργεια της Τουρκίας σημαίνει ότι τώρα ισχυροποιείται η Τουρκία και ε, συμμετέχει άμεσα στις εκαθαρίσεις ε, στα πεδία της μάχης. Θα πρέπει να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση μιας πραγματικά πολιτικής ένωσης. Ευχαριστώ. Περνούμε τώρα στη διαδικασία του Catch the Eye. Ε, μπορείτε να ζητήσετε το λόγο βάσει του άρθρου 16. Ε, πρώτα, κυρία Ρόζεμπεργκ, ένα λεπτό. Η Τουρκία για μια ακόμη φορά υλοποιεί τα παράνομα σχέδιά της περιφρονώντας το διεθνές δίκαιο εισέβαλε στη βόρεια συρία σκορπώντας θάνατο εκτοπισμό χιλιάδων και προσφυγιά. επιχειρεί εθνοκάθαρση με ευρωπαϊκά κονδύλια εγκληματώντα κατά της ανθρωπότητας. οι ηνωμένε πολιτείε η ρωσία ο ασαντ μετρούν κέρδη και ζημιές ενώ η δύση εμφανίζεται σε ρόλο αμήχανου παρατηρητή. οι αξίες μας κλονίζονται και έχουμε ευθύνη γι' αυτό συνάδελφοι διαχρονικά η τουρκική πολιτική του αναθεωρητισμού δεν έχει αρχές δεν σέβεται διεθνείς κανόνες και δεν υπολογίζει κανένα. πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα σε υλοποίηση στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων με σεβασμό στην κοινωνία των πολιτών και να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα στην τουρκία ότι με δική της ευθύνη δεν είναι ευπρόσδεκτη στην ευρωπαϊκή οικογένεια. σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μαυρίδης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Διαβάζω τον τίτλο «Η τουρκική επιχείρηση στη βορειοανατολική Συρία και οι συνέπειες». Θα ήταν καλύτερα να πούμε ότι δεν πρόκειται μόνο για στρατιωτική επιχείρηση. Πρόκειται για στρατιωτική εισβολή και οι επιπτώσεις δεν αφορούν μόνο την ασφάλεια ε, ή την προδοσία των Κούρδων ε, συμμάχων ε, και την ισχυροποίηση της μάστιγας του, του ISIS. Πρόκειται για συγκεκριμένα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εθνοκάθαρση δηλαδή και σχέδια για παράνομους ε, στη Συρία. Ε, αυτό μας θυμίζει την ε, εισβολή στην Κύπρο. Όπως το Αφρίν, ε, μετά το Αφρίν μπορούμε να συντρίψουμε την οικονομία του Ερντογκάν. Μπορούμε να λάβουμε άλλα μέτρα, μπορούμε να φέρουμε τους εγκληματίες στη δικαιοσύνη. Ήρθε η ώρα γι' αυτό. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπιλμπάου Μπαραντίκα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω την πλήρη μας απόρριψη στην παράνομη εισβολή της Τουρκίας. Αυτή η εισβολή παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δημιουργεί ε, θύματα μεταξύ των πολιτών. Επίσης ζητά να αλλοιώσει την παρούσα δημογραφία και να, και να εγκαταστήσει 3,5 εκατομμύρια ε, πρόσφυγες σε μια περιοχή που έχει εντελώς διαφορετική σύνθεση πληθυσμού. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται συγκρούσει τι οποίε ενέχονται όλες οι παγκόσμιες ε, δυνάμεις. Τα Ηνωμένα Έθνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καταπολεμήσουν αυτή την κατάφορη παραβίαση του διεθνού δικαίου με την επιβολή ουσιαστικών ε, κυρώσεων. Θα πρέπει να βρεθεί μια λύση σε διπλωματικό επίπεδο, η οποία να συνδυαστεί με την παροχή ανθρωπιστική βοήθεια, ε, φυσώντας την περιοχή, ε, φυσώντας την παγκόσμια προσοχή στην ε, ευάλωτη αυτή περιοχή της Συρίας. Ευχαριστούμε κυρία Κάμπα για ένα λεπτό. Ε, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. έχουμε αναπτύξει στο επίπεδο της ε, διπλωματίας αποτελεσματικά εργαλεία. Και τι γίνεται τώρα. Η Ρωσία βρίσκεται μπροστά μας και έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι ημών και αυτό είναι εξαιρετικά θλιβερό. Η Ευρώπη πάσχει ε, από τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στην Αγγής Ανατολή. Γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας ούτως ώστε να τερματιστεί αυτή η σύγκρουση όχι μόνο σε ελεκτικό επίπεδο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να πετύχουμε μια λύση σε διπλωματικό επίπεδο. Ε, θα πρέπει επίσης να φροντίσουμε για τα θύματα και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο κύριο Στυλιανίδη γιατί κάνει πολλά για τα θύματα. Ωστόσο, στην Αγγλική Ανατολή στη Συρία υπάρχουν επίση κάποιοι θελοντές οι οποίοι υποστηρίζουν τους πρόσφυγες εν μέσω πολλών κινδύνων. Οι οργανισμοί αυτοί θα έπρεπε να υποστηριχθούν. Επόμενο ο ο κύριος Παπαδημούλης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Λόγια, λόγια, λόγια. Ο Ερντογάν εισβάλλει στη Συρία με πράσινο φως από τον τραμπ με τις πλάτες του πούτιν κλείνουν συμφωνίες σε βάρος του διεθνούς δικαίου και της νομιμότητας αναθεωρεί τη συνθήκη της λοζάνης και η ευρωπαϊκή ένωση στην πράξη αποδεικνύεται ένας πολιτικός νάνος διότι δεν αρκούν τα λόγια της καταδίκης χρειάζονται έργα στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις αποτελεσματικό εμπάργκο όπλων υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση του συμβουλίου εδώ και μερικούς μήνες στην οποία συνέβαλαν ο αλέξης τσίπρας και ο πρόεδρος αναστασιάδης. είναι ώρα να εξειδικευτεί και να εφαρμοστεί και αυτό δυστυχώς το εμποδίζουν για κοινικά οικονομικά συμφέροντα κυβερνήσεις όπως της γερμανίας και της γαλλίας. ας είμαστε ειλικρινεί. Thank you, Madam One minute. Κυρία Σιόιντροβα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Θα πρέπει να καταδικάσουμε την τουρκική εισβολή στη Συρία. Η επίθεση αυτή ήταν εις βάρος και εναντίον αυτών οι οποίοι πολέμησαν το Ισλαμικό κράτος. Η παρέμβαση αυτή δυστυχώς δημιουργεί αστάθεια, νέα κύματα προσφύγων και δυστυχώς επίσης και κυρίως απώλειες ανθρώπινης ζωής, απώλειες αθώων. Είναι θετικό τουλάχιστον το ότι η Τουρκία έχει διακόψει την επίθεσή της ε, μετά από πίεση από τη ΣΥΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια ζώνη ασφαλείας στη Βόρεια Συρία θα μπορούσε να έχει μόνιμα ε, σημασία ε, αν ήταν δυνατόν να ελέγχεται από διεθνείς δυνάμεις και όχι από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Το τελευταία χρόνια η Τουρκία γενικά συμπεριφέρεται σαν χώρα που δεν σέβεται καθόλου τις ευρωπαϊκές αξίες. Η κυρία Ward. Εκατομμύρια κάτοικοι διαφορετικών εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων απειλούνται. Ε, δεκάδες χιλιάδες έχουν ουσιαστικά εκτοπιστεί. Ε, κουρδικά χωριά, χριστιανικές γειτονιές στις Συριακές πόλεις έχουν γίνει στόχος βολών ε, των επιτιθέμενων. Προκαλούνται δημοκρατικές αλλοιώσεις και αλλαγές Εγώ έχω επανειλημμένα πει ότι θα πρέπει να σταματήσει αμέσως η εισβολή και κατοχή των Τούρκων στη Βόρεια Συρία. Και θα πρέπει να δημιουργηθεί μια περιοχή ασφαλής, θα πρέπει να σταματήσουν τα όπλα να σειραίουν στην Τουρκία και να προλάβουμε περαιτέρω εγκλήματα και εθνικές εκαθαρίσεις από πλευράς είτε των Τούρκων είτε των, του ISIS. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να υπάρξει μια πολιτική λύση με τη συμμετοχή των γυναικών και όλων των θρησκευτικών και εθνοτικών κοινοτήτων. Γιοβέβα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Υποστηρίζω το ψήφισμα αυτό. Συμφωνώ με την έκλαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις πιστώσεις της Ευρωπαϊκές που δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ε, για την χρηματοδότηση στρατιωτικών επιχειρήσεων και δεν θα πρέπει να επιτρέπουν ε, στον Ερντογάν να μας εκβιάζει και δεν θα πρέπει οι τρίτες χώρες να παρεμβαίνουν στην περιοχή δεν θα πρέπει να υπάρχουν ε, ε, θάνατοι αθών και τέτοιου είδους καταστροφές. και απαιτείται να υπάρξει ουσιαστικό ευρωπαϊκό εμπάργο στα στρατιωτικά μέσα και να υπάρξει και μία ζώνη απαγόρευσης ε, υπέρτησης. Ε, υποτίθεται ότι τώρα πια η Τουρκία σταμάτησε μετά από πιέσει την επίθεση. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος της περιοχής εξακολουθεί να ζει κάτω από τον φόβο. Απαιτείται μια κοινή λοιπόν πολιτική και να αναλάβουμε επιτέλους τον πολιτικό ρόλο που μας αναλογεί. Σας ευχαριστώ. Οι στρατιωτικές επεμβάσεις στη Συρία είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και 7-8 χρόνια ε, υπεύθυνοι είναι χώρες όπως οι Ηνωμένε Πολιτείες που σε συνεργασία με χώρες συμμάχους όπως η Τουρκία, το Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Κατάρ εξόπλισαν στρατιωτικές δυνάμεις που είναι υπεύθυνε για δεκάδες χιλιάδες νεκρούς στην περιοχή κάτι το οποίο κατέστρεψε πολιτιστικά, κοινωνικά και οικονομικά την συγκεκριμένη χώρα. Οι ευθύνες λοιπόν που έχουν και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μεγάλες και οι αντιδράσεις που προέρχονται από πλευράς της είναι υποκριτικές και έτσι και αλλιώς ανεπαρκέστατες. Πρέπει να βοηθήσουμε την ανεξαρτησία και την εθνική και εδαφική ακεραιότητα της Συρίας σύμφωνα με, τους, ε, με τις ρυθμίσεις και τους κανονισμούς της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να θυμίσω ότι πέρα από την επίθεση ε, στη Συρία αυτό το οποίο, αυτοί οι οποίοι υποφέρουν ε, περισσότερο είναι τα παιδιά. Ε, τα παιδιά και οι ανήλικοι είναι αυτοί οι οποίοι υποφέρουν από, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο σε πολεμικές ε, συγκρούσεις. 70.000 είναι τα παιδιά που έχουν ε, αναγκαστεί να μείνουν μόνα τους και να φύγουν από τότε που ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες και που είχαν πάντα και έχουν ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας. 30 ε, χρόνια έχουν περάσει από τότε τα Ηνωμένα Έθνη και εμείς ρίξαμε την διακήρυξη για τα δικαιώματα των παιδιών. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι έτσι ώστε να δώσουμε τις μέγιστες δυνατές εγγυήσει στα παιδιά που παρά τη βούλησή τους έχουν εμπλακεί σε αυτή την ένοπλη σύγκρουση. Wallace, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Τουρκία πέρασε τα σύνορα και μπήκε στο κυρίαρχο κράτος της Συρίας. Παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Εισέβαλε στη Συρία, όχι στο Κουρδιστάν. Πρέπει να εκφράσουμε αλληλεγγύη προς τους Κούρδους. Αλλά η εδαφική κυριαρχία της Συρίας πρέπει να προστατευτεί από, από την ε, Συρία. Στην ε, Τουρκία ζουν πολλοί ε, Σύριοι που αντιμετωπίζονται ε, Η Τουρκία πήγε να πολεμήσει τους ε, ε, αντάρτες. Όταν επιστρέψουν στην Τουρκία όμως αυτοί ονομάζονται τρομοκράτες. Η Ευρωπή έδωσε 6 τα τελευταία δύο χρόνια στην Τουρκία για να αποτρέψει να κρατήσει τις, ε, τους πρόσφυγες που καταστράφηκαν τα σπίτια τους να μην έρθουν στην Ευρώπη. Ε, πώς επιτρέπουμε να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Η κυρία Γκραπίνη, τελευταία ομιλήτρια, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, έχετε τη δυνατότητα εδώ να παρατηρήσετε ομοφωνία στο Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο, η Επιτροπή επέκριναν αυτήν την επίθεση, αυτήν την εισβολή της Τουρκίας στη Συρία. Η κριτική δεν αρκεί όμως. Υπάρχει ένα ψήφισμα, θα ψηφιστεί αύριο, αρκεί όμως αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με άλλα θεσμικά όργανα υποχρεούται να παρέμβει με συγκεκριμένα μέτρα. Τι μπορούμε να κάνουμε. Η Τουρκία είναι σημαντική, είναι σημαντική και ως αγορά. Αλλά τι θα επιλέξουμε να κάνουμε να αναπτύξουμε την εσωτερική αγορά και την οικονομία ή να φροντίσουμε για την ασφάλεια των ανθρώπων που πεθαίνουν εκεί. Γυναίκες, παιδιά, άνθρωποι που πρέπει να τους προστατέψουμε, γιατί ένας στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την ειρήνη και την ασφάλεια. Και όπως έλεγε και χθε ο κύριος Γιούγκερ, εμείς έχουμε ειρήνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αρκεί αυτό. Έχουμε και διεθνή ευθύνη και πρέπει να κάνουμε περισσότερα πέρα από ένα ψήφισμα. Ευχαριστώ. Η κυρία του για ε, την ύπατη εκπρόσωπο της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Έχετε το λόγο. Αυτή η συζήτηση ήταν πολύ χρήσιμη και επίκαιρη. Με αυτή την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω τα αξιότιμα μέλη για τις παρεμβάσεις τους, τα σχόλια και τις προτάσεις τους. Η τουρκική μονόπλευρη επέμβαση στη Συρία προκάλεσε και εξακολουθεί να προκαλεί τεράστια ανθρώπινα δεινά, υπονομεύει την ε, μάχη κατά του ISIS, απειλεί την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Για όλους αυτούς τους λόγους, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και πάλι την Παρασκευή εκάλεσε την Τουρκία να τερματίσει τη στρατιωτική επιχείρηση, να αποσύρει τις δυνάμεις της και να ε, σεβαστεί το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Το Ευρωπαϊκό ε, συμβούλιο ε, θα ε, συνεχίσει να παρακολουθεί το θέμα. Επίσης, αντιμετωπίζει την ανθρωπιστική κρίση με βάση τις ανάγκες. Επιμένουμε σε μία πλήρη πρόσβαση των εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις για να βοηθήσουν όσους υποφέρουν επί τόπου. Η προστασία των αμάχων θα πρέπει να παραμείνει απόλυτη προτεραιότητα. Τώρα, σχετικά με τη λεγόμενη συμφωνία στο Σότσι χθε για την αποκλιμάκωση των επιχειρήσεων. Ελπίζομαι ότι θα σώσει ζωές και θα προλάβει περαιτέρω δυνάτων αμάχων. Ως προς αυτό ότι χαιρετίζομαι ως προσπάθεια να ε, σταματήσει τον κύκλο της βίας. Θα πρέπει να δούμε ε, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι επιπτώσεις θα έχει αυτή η συμφωνία στο Σότσι. Ένα πράγμα δεν άλλαξε όμως. Αυτό που χρειάζεται για να σταματήσει σε μόνιμη βάση η διένεξη στη Συρία είναι μια συνολική συμφωνία για τη Συρία που θα διαπραγματευτούν οι Σύροι για τους Σύρους ε, παράλληλα με το ψήφισμα 2254, ε, το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών. Μέχρι τέλος του μήνα θα, φτάσει, θα συζητηθεί στη Γενέβη το θέμα και μετά ε, ελπίζομαι ότι θα οικοδομηθεί μια μόνιμη λύση. Θέλω να εκφράσω την εκτίμησή μου για τη συνεχή σας προσπάθεια να εξευρεθεί μια διαρκής και μόνιμη λύση ε, στην σύγκρουση αυτή στη Συρία. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ ε, και τον Επίτροπο Στυλιανίδη που παρέμεινε και παρακολούθησε τη συζήτηση. Η συζήτηση κλείνει, θα ψηφίσουμε επί ενός ε, ψηφίσματος. Έχουμε 7 προτάσεις ψηφίσματος. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Οι ψηφοφορίες θα ακολουθήσουν σε λίγο. Ευχαριστώ. Herr President. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Λοιπόν, άρχεται η συνεδρίαση. Παρακαλώ να καθίσετε. Ich darf Ihnen bekannt geben. Θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω όσον αφορά την ε, ε, εκλογή του διαμεσολαβητή στις 16 Σεπτεμβρίου ενημερωθήκατε για τις εκλογές αυτές. Μέχρι τις 30 ε, Σεπτεμβρίου έχουν φτάσει πέντε ε, πέντε υποψηφιότητε, οι οποίε ε, εγκρίθηκαν όλες. Οι υποψήφοι είναι ο κύριος Γκουτζέπε Φορτουνάτο, η κυρία Τζούλια Λαφράνκ, ο κύριος Νίλς Μουίσνικ, η κυρία Έμιλι Ορέιλι και η κυρία Σεσίλια Βίξτραμ. Ε, στοιχεία για του υποψηφίου.